πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου. Και τώρα προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, που αφορά το Πεκίνο 15 χρόνια μετά προφορική ερώτηση της κυρίας Εύαν Σφένσον για τη θέση της ε, γυναίκας και την ισότητα μεταξύ των φίλων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Τα θέματα των γυναικείων δικαιωμάτων ήταν ανέκαθεν προτεραιότητα για μένα προσωπικά και γι' αυτό και χαίρομαι που ε, είναι προς σήμερα προσυζήτηση εδώ στην Ολομέλεια. Στην Επιτροπή των Γυναικών υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα που αντιπροσωπεύει τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πλατφόρμα του Πεκίνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής αυτής που συνεργάστηκαν τόσο καλά μεταξύ τους και μαζί μου. Η υιοθέτηση της πλατφόρμας το 1995 από τον ΙΕ ήταν ένα ιστορική σημασίας βήμα. Η πλατφόρμα για δράση, όπως αποκαλείται, ήταν το πρώτο τέτοιο είδους έγγραφο. Και κρατούσε μία ε, αποτελούσε μάλλον μια γενική εικόνα, μια γενική άποψη για την θέση της γυναίκας στην Ευρώπη. Μόνο το 1948 θα πρέπει να θυμηθούμε ότι οθετήθηκε η καθολική δήλωση, διακήρυξη μάλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, αυτή η διακήρυξη συμπεριλαμβάνει 30 άρθρα και πολύ συχνά αναφέρονται και εκεί, στο δεύτερο άρθρο λοιπόν, λέει συγκεκριμένα ότι τα δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει να προστατεύονται. Εντός της Ένωση, το θέμα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί, έχει μάλλον βάση νομική τόσο στις συνθήκες όσο και στο χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Επιτροπή είμαστε σύμφωνοι για τη σημασία της πλατφόρμας του Πεκίνου και την ανάγκη να συνεργαστούμε και να εργαστούμε μάλλον αντωνότερα ώστε να οθήσουμε τις εξελίξεις και να διασφαλίσουμε την ε, εξέλιξη προς μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει στο Βίλνιους να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις τελευταίες έρευνες και τις πιο αποτελεσματικές ε, και να προσπαθήσουμε να βρούμε τις πιο αποτελεσματικές πολιτικές λύσεις. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δεν έχουμε και εγώ στηρίζω την πρόταση για ε, ένα ευρωπαϊκό ε, διάταγμα προστασία που πρότεινε η Ισπανική Προεδρία. Στην πλατφόρμα του Πεκίνου υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία είναι πολύ κρίσιμα για να μπορέσουμε να, αν θέλουμε να πετύχουμε. Φτώχεια που επηρεάζει τις γυναίκες πολύ δυσανάλογα, η άνηση πρόσβαση στην ε, υγειονομική περίθαλψη, η βία κατά των γυναικών που παίρνει πολλές μορφές, ανισότητα στις οικονομικές δομές και στην οικονομική πολιτική. Όπως γνωρίζετε, μια αντιπροσωπεία 8 βουλευτών θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να εκπροσωπήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση και τις διαπραγματεύσεις που θα αποτελέσουν ακόμα ένα βήμα προς την αξιολόγηση για το πόσο έχουμε προχωρήσει τα τελευταία 15 χρόνια ώστε να εκπληρώσουμε τους στόχους ε, της ε, πλατφόρμας και το ψήφισμα που θα υιοθετηθεί αύριο θα είναι αυτό που θα πάρουμε μαζί μας ε, στις βαλίτσες μας για τη Νέα Υόρκη. Στην Επιτροπή υιοθετήσαμε επίσης και το δικαίωμα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής ζωής και αυτό είναι μέρος των γυναικείων δικαιωμάτων και θα πρέπει να βελτιωθεί στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε αυτό το σημείο να ψηφιστεί χωριστά. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ε, ζητείτε χωριστή ψηφοφορία για ένα σημείο είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο και γι' αυτό και δεν θα ψηφιστεί αν μπλοκ με το υπόλοιπο του ψηφίσματος. Εγώ συμφωνώ με το ΕΛΚΟ πως ε, αυτό το κομμάτι, το τμήμα 9, είναι, η παράγραφος 9 είναι μεγάλη σημασία, αλλά έχω την εντύπωση πως θέλουν να καταψηφίσουν την παράγραφο αυτό και πιστεύω πως θα ήταν πραγματικά κρίμα. Γνωρίζω πολύ καλά πως εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε διαφορετικές απόψεις και αξίες, όμως ε, ε, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε συζήτηση, γίνεται συζήτηση. Το κείμενο αυτό όμως είναι, ένα, είναι κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές και πιστεύω πως όλοι θα μπορούσαν να τις υποστηρίξουν και δεν είχε προταθεί άλλο κείμενο για την κατάσταση της της παραγράφου 9 και θα ήταν κρίμα να φτάσουμε σε ένα ψήφισμα που να μην λέει ούτε καν το αμήνυμο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα κλειδί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω και ελπίζω πως όλοι θα μπορέσετε να δεχτείτε το κείμενο ως έχει, διότι λέει πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα για όλους μας. Και σε αυτή τη διαδικασία έχουμε συνεργαστεί στενά με χιλιάδες ε, οργανώσεις γυναικών και τα μέλη τους. Το έγγραφο αυτό πραγματικά έχει ευρύτατη βάση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωπος του Συμβουλίου, Λόπες Γαρίδο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Σβέντσον. Επίσης, ευχαριστώ για την ερώτησή σας, κυρία μου, διότι θα γνωρίζετε ότι η Ισπανική Προεδρία θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ βασικό θέμα η ισότητα. Και το έχουμε τάξει αυτό ως στόχο της πολιτικής μας. Γι' αυτό και προωθούμε την οδηγία κατά των δυσμένων διακρίσεων και όπως και εσείς είπατε. Θεωρούμε ότι είναι βασικό να καταπολεμήσουμε την βία μεταξύ των δύο φίλων και να προστατεύσουμε τα θύματα της. Και επίσης ε, συνεργαζόμαστε και με την ε, Επίτροπη κυρία Ρέντινγκ που στο χαρτοφυλακιό της έχει και αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, λοιπόν, θα που δεν μπορείς να παραστεί εδώ η Υπουργό Ισότητα τη ε, κυβέρνησή μα, διότι έπρεπε να παραστεί στη Γερουσία σε σχέση με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις αμβλώσεις. Ε, ήδη εγκρίθηκε το σχετικό νομοθέτημα στην Βουλή της χώρας μας. Ανέκαθεν ασπαζόμασταν τα όσα πρεσβεύει ο ΙΕ για την ισότητα και συμμετέχουμε και στην αντίστοιχη επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών, οπότε και εμείς αναδεικνύουμε ως προτεραιότητα το ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας όσον αφορά την πλατφόρμα του Πεκίνου. Όπω τα γνωρίζετε, έχουμε κάνει κάποια βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Απάντω, ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλαμε. Και γι' αυτό και πρόκειται και τον Μάιο να έχουμε μια εκδήλωση, ούτως ώστε να συζητηθεί το τι γίνεται με τα στερεότυπα σε σχέση με την ισότητα των φύλων στα ΜΜΕ. Και εκεί βεβαίω θα συμμετάσχει η αρμόδια επιτροπή κ. Βιβιαν Ρέντι. Εν κατακλείδη θέλουμε να σας πούμε ότι υπάρχει ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που γνωρίζετε όλοι. Πρόκειται για την χρηματοπιστωτική κρίση. Διότι πέραν των άλλων ε, κακών συνεπειών Άλλη αρνητική συνέπεια είναι και ότι αποτελεί φραγμό και για την πρόοδο στην ισότητα ανδρών και γυναικών. Όμω από την άλλη μεριά, κατά τρόπο παράδοξο, μπορεί να μα βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση η ισότητα και για παράδειγμα η ισότητα στην πρόσβαση στη δουλειά. Να σας παραπέμπω και στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, όπου είναι ξεκάθαρο ότι η στρατηγική του 2020 πρέπει να έχει, είπαμε, μία τέτοια εγκάρσια διάσταση που να αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχετική έκθεση πέρσι ζήτησε από Κομισιόν και Συμβούλιο να έχουν ειδικό κεφάλαιο στην στρατηγική του 2020. Στις 30 Ενδεκάτου το Συμβούλιο στην ε, Βαρκελόνη κατέληξε στο ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους να μπορέσουν αυτή τη διάσταση, τη διάσταση της ισότητας να την ενσωματώσουν στην πολιτική για την Ευρώπη του 2020. Αυτό είναι κάτι που να καλύψει όλες τις πολιτικές πτέρυγες. Να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα εργασίας που πάντοτε ήταν θεμέλιο για τέτοιες στρατηγικές. Είμαι δε βέβαιος ότι το έγγραφο το οποίο μας υποσχέθηκε να παρουσιάσει η Κομισιόν στις 3 Τρίτου για τη στρατηγική του 2020, όπως και σήμερα μας ε, είπε ο κ. Μπαρός, ο κ. Φενεροπάη, ότι και αυτό το έγγραφο λέγω πρόκειται να θίξει και το πρόβλημα που τώρα συζητούμε. Δεν είναι θέμα δικαιοσύνη μόνο, είναι θέμα συνέπειας με το πνεύμα που διαπνέει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε πάντοτε να σημείο αναφορά σε αυτή η ισότητα πάντοτε στον κόσμο. Η ισότητα ανδρών και γυναικών. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και καλώς ορίσατε κυρία Επίτροπε. Έχετε τις κοιτάλησεις. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, είναι τιμή που η πρώτη μου παρέμβαση ενώπιον του Κοινοβουλίου αφορά μια απάντηση θέματα γυναίκα. γιατί ως ε, επίτροπος αρμόδια για τα βασικά δικαιώματα νομίζω ότι το βασικό δικαίωμα της ισότητας ε, ε, μεταξύ των γυναικών είναι ένα από τα πιο παλιά και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ και 15 χρόνια ως νέα βουλευτής ε, από το Λουξεμβούργο προετοίμασα την πλατφόρμα για το Πεκίνο και τώρα εμείς εξετάζουμε εδώ τη συνέχεια της ε, πλατφόρμας αυτής του Πεκίνου. Κρίνες κύκλες λοιπόν. Δεν χρειάζεται να τονίσω, γιατί το ξέρετε, η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι μία από τις βασικές και ουσιαστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορείτε πραγματικά να βασιστείτε σε δέσμευση χωρίς σφάλμα της Κομισιόν σε αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντο έτο θα υποβάλω μια νέα στρατηγική τη Κομισιόν για θέματα ισότητα ανδρών και γυναικών που θα συνεχίσει αυτό που αναφέρεται στο φιλοπορίας για την ισότητα 2006-2010. Επίσης, το καθεστώς της γυναίκας ε, στα Ηνωμένα Έθνη που γιορτάζουν επίσης την 15η ε, επέτειο του Πεκίνου και εκεί θα αποστείλει σημαντική αντιπροσωπεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα είμαι παρόουσα μαζί με την πρόεδρο του Συμβουλίου και θα πρόκειται για μια πρεμιέρα γιατί και οι δύο θα μιλήσουμε στην ολομέλεια της συνάντησης αυτής και αυτό νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό σύμβολο. Επίσης θα είναι αυτή η σωστή στιγμή για να δούμε σε διεθνές επίπεδο ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στους 12 τομείς δράσεις που αναφέρονται στο Πεκίνο. Ακόμα και όταν δούμε ότι σε κάποιους τομείς εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα. Γιατί ακόμα και αν υπάρχει επιτυχία εν μέρη υπάρχουν ακόμα ανοιχτές προκλήσεις. Και θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θα παραμείνει ένας έντονος υποστηρικτής ε, των Ηνωμένων Εθνών και όσον αφορά τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να λάβουν χώρα τη δημιουργία αυτή της μονάδας ε, για το φύλλο επίσης στο ιστορικό των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Στηρίζει επίσης το θέμα της ανάπτυξης, ιδίως μέσα στα πλαίσια του στόχου της χιλιετίας, που εξασφάλουν μία σημαντική θέση. όπου οι πολίτες ανά τον κόσμο ξέρουν ότι χωρίς ισότητα των φύλων δεν θα υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια πολιτική οριζόντια ε, και θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική από την υπεύθυνη επίτροπο και από τους άλλους όλους επιτρόπους. Και υπάρχει αυτή η ευθύνη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όσον αφορά τις εξωτερικές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά την πολιτική συνεργασίας. Ξέρουμε όλοι ότι η εφαρμογή της πλατφόρμας δράσης ε, του Πεκίνου ήταν ένα σημαντικό βήμα και κατόπιν της υιοθέτησης πλατφόρμας αυτής μάλιστα γενικοποιήθηκε η ε, κάθετη συμπερίληψη του παράγοντα φύλλο σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Αυτό ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα του Πεκίνου τότε και οι επιπτώσεις ήταν σημαντικές γιατί σε όλα τα κράτη-μέλη η πολιτική ισότητα δεν περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες δράσεις αλλά έχει γενικευθεί σε όλες τις ε, αποφάσεις και τους νόμους. Η πολιτική αυτή βασίζεται σε δείκτες που αναπτύχθηκαν από το Συμβούλιο για τους περισσότερους τομείς δράσης. 12 δράσεις και 9 δείκτες υπάρχουν Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι λοιπόν για τα αποτελέσματα. Αλλά υπάρχουν και τρεις δείχτες που θα πρέπει ακόμα να δημιουργηθούν και νομίζω ότι αυτή είναι μια δέσμευση που πήρε το Συμβούλιο υιοθετώντα τα συμπεράσματά του για να μπορέσει να προχωρήσει και να αναπτύξει αυτούς τους δείκτες που λείπουν. 15η επέτειος της πλατφόρμας του Πεκίνου η Σουηδική Προεδρία πραγματοποίησε έναν απολογισμό. Το Συμβούλιο εθέτησε τα συμπεράσματα και το Κοινοβούλιο θα παρουσιάσει τα δικά του έγγραφα. Έγγραφα τα οποία σίγουρα θα βρουν τη θέση τους σε όλες τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η κυρία Πρόεδρος και ο κύριος Πρόεδρος αναφέρθηκαν στην Ευρώπη του 2020 είναι προφανές ότι το σύστημα αυτό που θα ξαναξεκινήσει την ανάκαμψη στην Ευρώπη έχει ένα σημαντικό ρόλο, ιδίως αυτή τη στιγμή που όσο πάει και περισσότερους εργαζόμενους χάνουμε και χρειαζόμαστε άρα τις γυναίκες για να μπορέσουν να υπομισθούν την οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο θέμα θεωρητικής ισότητας, είναι θέμα οικονομικής πολιτικής. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία επιλογή. Χρειαζόμαστε τις γυναίκες αν θέλουμε να βγει η Ευρώπη από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Και αυτοί οι νέοι δίχτες θα μας βοηθήσουν βέβαια και μέσα στα πλαίσια της ομάδας υψηλού επίπεδου προετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα εργασίας που θα μας επιτρέψει να δούμε τη συνέχεια για τους υπάρχοντες συντελεστές και να υιοθετήσουμε τους συντελεστές που θα πρέπει ακόμα να υιοθετηθούν. Και βέβαια εδώ θα μας βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Ανδρών και Γυναικών που ήδη την επόμενη εβδομάδα, γιατί και αυτό είναι ένα σύμβολο, στην δηλαδή που υπάρχει διάσκεψη στη Νέα Υόρκη, θα υπάρχει οριστική εγκατηθίδρυση στο Βίλνιους του Ινστιτούτου μας. Κύριε Πρόεδρε, σύντομα θα έρθω εδώ σε εσά μετά τη Νέα Υόρκη για να συζητήσω την στρατηγική της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα θέματα ισότητας. Θα το πετύχουμε αυτό από κοινού για όφελος του 50% του πληθυσμού, 50% των πολίτων και θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό που θα πετύχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, προς την Επίτροπο. Αναλαμβάνω και πάλι, όπω βλέπετε, την ε, Προεδρία. Θα συνεχίσω στα Ουγγρικά και επίση. Καλησπέρα, κύριε Επίτροπο, καλησπέρα, κύριε Γαρίδα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τώρα για την ισότητα των φίλων θα λάβουν το λόγο γυναίκε και οι 14 που είναι το λόγο είναι γυναίκε πρώτη-πρώτη, κυρία Κρίστα Κλά. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Οπωσδήποτε κάτι έχουμε να συμβάλλουμε. Αγαπητέ κυρία Πρόεδρε, η και η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών στην επόμενη εβδομάδα στην Νέα Υόρκη μα δίνει δυνατότητα να εστιάσουμε την προσοχή παγκόσμια στην ισότητα ανδρών και γυναικών. Και θα πρέπει εκεί με κριτικό πνεύμα να εξετάσουμε τι έχουμε πετύχει και τι θέλουμε ακόμα να πετύχουμε. Η πρόσκληση της Διεθνούς Διάσκεψης Γυναικών το 1995 στο Πεκίνο για ισότητα και ειρήνη εξακολουθεί να είναι ένα συγκεκριμένο στόχος για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προχωρήσουμε έχοντας πάντα κατά νου αυτό το στόχο. Ξέρουμε βέβαια ότι ο στόχος δεν είναι εύκολος, ότι σταματάμε, υπάρχουν μονόδρομοι. Θα πρέπει να το λύσουμε τα πράγματα πολύ καλύτερα και να έχουμε το θέμα πάντα κατά νου. λέμε ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη. Θα πρέπει να δούμε πού είναι τα κοινά σημεία. Η πολιτική ισότητα δεν μπορεί να είναι θέμα πλειοψηφία και ψηφοφορία. Η ομάδα μου αφήνει την ελευθερία για την ψηφοφορία. Γι' αυτό κυρία Σφένσον υπάρχει κατά τμήματα ψηφοφορία. Χρειαζόμαστε ε, ο καθένας να καταλάβει τι γίνεται η κυρία Σφένσον έθεσε το δάχτυλο από τον τύπο των ήλων πολλές φορές. Πολλά πρέπει να γίνουν, να μην είμαστε τυποποιημένοι στις σκέψεις μας, η βία κατά των γυναικών, η συμπληρωμή για την ίδια εργασία, ε, πολλά θέματα πάρα πάρα πολύ σημαντικά που θέλουμε να τεθούν μέσω της, ε, του ψηφίσματος αυτό. Αλλά δεν αρκεί να λέμε μονάχα τι θέλουμε να πετύχουμε. Η ομάδα μου θέλει κάθε φορά που αναφέρουμε το θέμα της ισότητας να αντιμετωπίζουμε ισότιμα τους άντρες και τις γυναίκες, να τους αναφέρουμε και τους μεν και τους δε. Και ελπίζω στην ε, διάσκεψη συνέχειας του Πεκίνου θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε να βήμα προς τα μπροστά. Ευχαριστώ. Και τώρα για ένα λεπτό, ενάμεση λεπτό, ο Η κυρία Γκουρμάη, συγγνώμη. Αγαπητέ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. 15η επέτος από την ε, δημιουργία της πλατφόρμας του Πεκίνου. Θα πρέπει να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε αλλά και να αναζητήσουμε νέους τρόπους για να επιτύχουμε τους επιθυμητούς στόχους. Η αρχή ήταν αφαιρετική, το 1995 επετεύχθη γενική συνένεση, άνδρες, γυναίκες, νέοι, Η, από την, την οικονομική, την νομική, την κοινωνική. Η, όμως παρά τη συνένεση οι συνέπειες οι απτές ήταν λιγότερο προφανή σε πολλέ χώρε οι γυναίκε εξακολουθούν να μην χαίρουν όλων αυτών των δικαιωμάτων και πολύ συχνά η φτώχεια είναι γυναικεία. Ε, ακόμα και στι αναπτυγμένε χώρε εξακολουθούν να υπάρχουν και να συζητήσει σε σχέση με ορισμένα θέματα όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπροβλητικά δικαιώματα και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο δεν ακολουθεί αυτή την τάση και κρατά σταθερή θέση, και ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτή το βασικό δικαίωμα. Ε, δεν έχει τελειώσει λοιπόν η συζήτηση. Ο αγώνας ε, των γυναικών δεν έχει τελειώσει. Δεν μπορούν τα δικαιώματα να είναι αντικείμενο συμβιβασμού και γι' αυτό και στη Νέα Υόρκη σε λίγες μέρες θα πρέπει να αναζητήσουμε την εγγύηση της απόλυτης προστασίας των δικαιωμάτων αυτών. Εγώ προσωπικά θα το κάνω σύμφωνα με το σλόγγαν, το σώμα μου και τα δικαιώματά μου και το ίδιο θα κάνω για όλες τις γυναίκες του κόσμου. Πρόεδρε, επίτροπε, συνάδελφοι, θα πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή για να δούμε τι έγινε από τότε που είχαμε αυτή την, ε, την, την πλατφόρμα του που έγινε πριν από 15 μέρε. Τότε θα διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα επιδέχονται βελτίωση, γιατί ακόμα είμαστε μακριά από εκείνου του στόχου. Ε, ανισότητα συνεχίζεται παντού στον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν θέλουμε να σημειωθεί πρόοδο για αυτά τα θέματα, τότε θα πρέπει να υπάρξει και σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο ε, κάποιο είδου συγκρισιμότητα των δικτών για τα θέματα του Πεκίνου και να εξασφαλίσουμε ότι είναι ενημερωμένοι αυτοί οι στόχοι, τόσο ώστε να έχουμε μια κατάλληλη στρατηγική και στην Ευρώπη ακόμα. Ε, έχουμε να βελτιώσουμε πολλά, να δούμε τι είναι στην αγορά εργασία, οπότε και θα πρέπει ε, ό,τι κενό υπάρχει να το, να άρουμε, θα πρέπει να είναι και σε διευθυντικέ ε, θέσει και οι γυναίκε σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα. Να σταματήσουν τι διακρίσει γιατί όλα αυτά συνήθως οδηγούν τις γυναίκες σε περιθωριοποίηση, σε, σε φτώχεια, το οποίο όμως έχει, να κάνει τελικά και με την ψυχή και τη διανοητική τους κατάσταση, δυσμενείς διακρίσεις, που πολλές φορές ε, ε δεν, δεν, έχουν την, προστασία, την, προστασία, την σημασία που θα έπρεπε και επίση οι Ρωμά, οι γυναίκε Ρωμά, πολλέ φορέ υφίστανται πολύ χειρότερα από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη και για τι ηλικιωμένε γυναίκε. Το προσδοκιμό ζωή, η διαφορά μεταξύ άντρων και γυναικών. Βεβαίω είναι και θέμα ε, ε, οικονομικό, θέμα και κοινωνικό για τι ε, ανήπαντρε μόνε φτωχέ γυναίκε. Οπότε θα πρέπει να απευθύνω έκκληση, κυρία Επίτροπη, να κάνετε μια οδηγία για τη βία των γυναικών και θα σα στηρίξουμε όλε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Από το 2006 ο ΙΕ διαπίστωνε ότι τα πιο ευάλωτα και πιο φτωχά άτομα είναι τα πρώτα θύματα των κλιματικών αλλαγών. Οι γυναίκες όμως είναι αυτές που πλειοψηφούν σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Στην Μαύρη Αφρική για παράδειγμα, ενώ ήδη υπόκειται διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση και τον έλεγχο της γης, η αποψήλωση των καλλιεργήσιμων γεών που προκαλείται από την ξηρασία περιορίζει ακόμη περισσότερο τα προστοζήν. Το 2.200 από ό,τι 2.100 ε, μάλλον ε, μέγα, μέγα κομμάτι του πληθυσμού θα έχει φύγει από τις ε, περιοχές αυτές και είναι αυξημένο το επίπεδο απειλών κατά των γυναικών. Ωστόσο πρέπει να διαπιστώσουμε ότι εδώ και 15 χρόνια ούτε ένα νομοθετικό κείμενο που υιοθετήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του περιβάλλοντος δεν έχει συμπεριλάβει την διάσταση του φύλου και ζητώ εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη να ενσωματώσουν την προοπτική ισότητα ανδρών γυναικών σε όλες τις αναλύσεις αντίκτυπου, τι νομοθεσίε και τι πολιτικέ που αφορούν, αφορούν το περιβάλλον. Σα ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η Μαρίνα Διανακουδάκη. Μόλις πριν 200 χρόνια έλαβαν το δικαίωμα ψήφου οι γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αγώνας για τα γυναικεία δικαιώματα δεν είναι νέο φαινόμενο και θέλω να τιμήσω όλες τις γυναικείες οργανώσεις στον κόσμο που εξακολουθούν να αγωνίζονται για την ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Ε, οι γυναίκες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες στις επιλογές τους για τη σταδιοδρομία τους ή για την οικογένειά τους, να μπορούν να δουλεύουν σε παραδοσιακά αρσενικές ε, δουλειές, αλλά και να μένουν οι άντρες να φυλάνε τα παιδιά στο σπίτι. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να δοθούν οι δυνατότητες στις ε, γυναίκες. Εμείς ως συντηρητικοί πιστεύουμε στην επιλογή. Επιλογή θα πρέπει να έχουν και οι γυναίκες και στη συνέχεια και η ισότητα. Μήπω χωρίς την πρόθεση καθιστούμε τις γυναίκες λιγότερο αποσχολήσιμε ζητώντας από τις επιχειρήσεις να προσφέρουν δικαιώματα ενώ δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά ε, μέσα στο πρόβλημα. Μήπως ε, επίσης θεωρούμε λιγότερο σημαντική την ανασχόληση με τα παιδιά από την ε, εργασία στο χώρο εργασίας. Η Κομισιόν ζητά να βγουν οι γυναίκες από την ύφεση και να ξαναβρούν δουλειά. Εγώ λέω πως θα πρέπει να βρουν δουλειά και με μικρές επιχειρήσεις. Με την υπερβολική νομοθεσία οι μικρές επιχειρήσεις μπορεί να αναγκαστούν ε, να, να εξοντωθούν και έτσι να σπαταλήσουμε τους λιγοστούς πόρους που έχουμε να αφιερώσουμε στις γυναίκες και έτσι να μην φτάσουν στην ισότητα την οποία αξίζουν. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η Μάρα Μπιζότο για ένα λεπτά. Η έκθεση της Σουδικής Προεδρίας δεν κάνει καμιά αναφορά στην κατάσταση της γυναίκας στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα δεν υπάρχει το πρόβλημα ή δεν θέλουμε να το δούμε. Και όμως η κατάσταση των γυναικών της Ισλαμικής, στις χώρες Ισλαμικής κουλτούρας είναι ακόμα χειρότερη από ό,τι παλιότερα. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτά τα επιχειρήματα που είναι στην καρδιά των αγώνων πολλών μουσουλμάνων γυναικών ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα πρέπει να δεχτούμε τη νέα πρόκληση και να την αναλάβουμε. Οι Ευρωπαίες και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να υποστηρίξουν την ε, γυναίκα μουσουλμάνα στην Ευρώπη, να τη βοηθήσουν ε, και να βοηθήσουν εκείνα τα κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο που υψώνουν τη φωνή τους κατά του Ισλαμικού φανατισμού. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε γι' αυτό, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για την κατάσταση των ε, μουσουλμάνων γυναικών στην Ευρώπη. Το πνεύμα αντιπαράθεση, αν οδηγήσει στην ε, σιωπή, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε το αίτημα της απελευθέρωσης των γυναικών κατά της καταπίεσης του Ισλαμισμού. Σα ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μπάουερ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. 15 χρόνια μετά από την σύνταξη της πλατφόρμας του Πεκίνου έχουν συμβεί διάφορα πράγματα αξιόλογα θα μπορούσα να μιλήσω για αυτά. Ωστόσο, εγώ θα μιλήσω για τα του οίκου μας. Και κατά αυτά τα τελευταία 15 χρόνια στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη έγιναν κάποια βήματα προς τα εμπρός και πρώτα-πρώτα είχαμε την, ε, ε, ε, ε, νόμους που θεσπίστηκαν κατά της δυσμενούς διάκρισης οπότε όλα αυτά είναι ένα βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά το ότι δημιουργήθηκε μια κατάσταση η οποία παρέχει εγγυήσει ισότητας ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες όμως δεν είναι δυνατόν να είμαστε τόσο ικανοποιημένοι για το ότι ε, έχει προχωρήσει όσο έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε θέσπιση και άλλων νομοθετημάτων. Δεν είμαστε πάντα όσο αποτελεσματικοί θέλουμε, γιατί πολλές φορές περνάει ένας νόμος, αλλά ο νόμος αυτός δεν περνάει στην νοοτροπία. Να, ας πούμε για την μισθολογική ισότητα. Εδώ και 30 χρόνια έχουμε τέτοιου είδους, ε, τέτοιου νομοθεσίες. Παρ' όλα αυτά συνεχίζονται οι μισθολογικές ανισότητες. Και πολλές φορές παραξύνονται ακόμα περισσότερο διαφορέ. Επομένω, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την, την, την ε, δικαστική αρρωγή, γιατί πολλέ φορέ νομικέ συμβουλέ κοστίζουν. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα, θα προσέξουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση γιατί πολλές φορές θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να έχουν την πλαισίωση πόρους που χρειάζονται ε, δεν μπορεί να λάβουν δράση. Απλώ κάτι συμβολέ δίνουν και ενημερώνουν. Ε, ελπίζουμε ότι επομένω και φέτο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση για να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η νομοθεσία που περνάμε, που εγκρίνουμε, που θεσπίζουμε. Άρα θα πρέπει να δούμε πώ θα προχωρήσουμε ε, και στη αλλαγή του νοοτροπίας γιατί τα στερεότυπα δεν αλλάζουν με μόνο θέσπιση νομοθεσίας. Να γιατί δεν έχουμε πετύχει επίσης θα πρέπει να σκάτσουμε να κάνουμε μια καταγραφή του τι έγινε μέχρι σήμερα. Και μετά να ταινίσουμε το μέλλον και να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε γιατί σίγουρα και ε, πάρα πολλές ελπίδες ε, και προσδοκίες θα έχουμε όσον αφορά την, στρατηγική 2020. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η υπόθεση να λεφτεί υπόψη για αυτή την στρατηγική ο Επίτροπος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάβερ. Και τώρα η Εντίτ Εστρέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρία Επίτροπε, με μεγάλη μου χαρά ακούω ότι στέλνετε ένα θετικό μήνυμα, πολύ θετικό μήνυμα. Γιατί είπατε ότι έχετε την πολιτική βούληση να αναλάβετε δράση. Ξέρετε, χρειαζόμαστε την ανάληψη δράσης, διότι 15 χρόνια μετά από το Πεκίνο διαπιστώνεται ότι δυστυχώς οι επιδόσεις μας συνεχίζουν να είναι φτωχές. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν αλλάζει ε, το, το ότι η φτώχεια είναι θηλυκή. Εξακολουθούμε να έχουμε αναλφαβητισμό και χαμηλούς μισθούς. Υπάρχουν διακρίσεις στην πρόσβαση στην παιδεία και είναι γυναίκες θύματα βίας ψυχολογικής και φυσικής. Οι γυναίκες υπό αντιπροσωπεύονται και στην πολιτική και στις ε, επιχειρήσεις και στην ουσία δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων είτε οικονομικής φύσεως είτε πολιτικής φύσεως. Γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές ισότητας πρέπει να είναι αποτελεσματικές και θα πρέπει και η διάγνωση να είναι αξιόπιστη, να βασίζεται σε συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία και διαιρεμένα αναφύλο. Αυτό χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια σωστή διάγνωση και μετά να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Σας ευχαριστώ buenas noches. Quería decir que yo no he venido Θα ήθελα... Δεν ήρθα εδώ στο Κοινοβούλιο για να χειροκροτήσω τον Ισπανικό νόμο για την σε εκτρώσεις που μόλις υιοθετήθηκε γιατί εγώ θέλω να υποστηρίξω την ανθρώπινη ζωή. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω την ζωή των γυναικών των οποίων η ζωή απειλείται εξαιτία της βίας της οποίας είναι θύματα. Θέλουμε να έχουμε ένα ε, χώρο ασφάλειας το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ζητεί να υπάρχει μηδενική ανέχεια έναντι όλων των βιωτήτων κατά των γυναικών και να υιοθετηθούν τα απαραίτητα μέτρα για την κατάλληλη προστασία των θυμάτων. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης έχει ορίσει ασφάλεια μεταξύ των άλλων για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Και θα ήθελα η Ισπανική Προεδρία να προωθήσει τα θέματα ασφαλείας των γυναικών που είναι θέματα, θύματα βίας. Ο αγώνας κατά της βίας των φίλων στην Ευρώπη δεν πρέπει να έχει σύνορα. Ο αγώνας κατά της κακομεταχείρισης των γυναικών θα πρέπει να ξεπερνάει τα νομοθετικά εμπόδια. Τουλάχιστον μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύουμε τη ζωή των γυναικών και των παιδιών τους. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο να πράξουν τα απαραίτητα και ό,τι είναι ανθρώπινο για να μπορέσει να προχωρήσει το ευρωπαϊκός νόμος που θα καταπολεμά την ατιμορρησία αυτών που ασκούν βία κατά των γυναικών. Η κυρία Γκαρσία Πέρες. Πριν από 15 χρόνια 30.000 γυναίκες ένωναν τη φωνή τους για να προχωρήσουν σε μια κοινωνία πιο ενωμένη και πιο ίση. Ήταν ενωμένε ε, για την αναγνώριση των δικαιωμάτων ισότητας και δικαιοσύνης, για την κοινωνική και πολιτική προστασία των γυναικών, για την κατανομή ευθυνών, για την προστασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Αυτοί οι στόχοι εν μέρη μπορεί να έχουν εκπληρωθεί αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν θα πρέπει να συνεχίσει με το, με πρόγραμμα εργασίας και την πρόθεση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων μέσα από νομοθετικές διαδικασίες και μέτρα. Στόχος μας είναι η ισότητα, αλλά στην προσπάθειά μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε και όλες εκείνες τις γυναίκες που έξω από την Ευρώπη πλήττονται από την έλλειψη νομοθεσίας που να τις προστατεύει. Και για αυτές τις γυναίκες πρέπει να παλέψουμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι η Μαρία Μαρέλσενα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, σχετικά με το ψήφισμα αυτό για ε, την το συνέδριο του ΟΗΕ για την ισότητα των ανδρών και γυναικών σκέφτομαι εδώ στο θέμα της απασχόλησης όπου οι διαφορές της αμοιβή είναι πολύ σημαντικές και πρέπει ακόμη να καθοριστεί το οικογενειακό πλαίσιο και βλέπω πολλά θέματα παρόλα στις ανισότητες όλες οι δράσεις του Πεκίνου 15 δεν έχουν ολοκληρωθεί και ε, γνωρίζουμε μεν καλά τους στόχους μας αλλά πρέπει πρέπει να εξετάσουμε ποιους τρόπους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να τους υλοποιήσουμε διότι αναφερόμαστε στο πρόγραμμα δράσης ε, των Ηνωμένων Εθνών σε τρεις άξονες καταρχήν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα βραχυπρόθεσμα να εξετάσουμε όλα τα ευαίσθηκα θέματα που επηρεάζονται από την οικονομική κρίση να έχουμε συγκεκριμένους δείκτες για να μετρήσουμε την επίπτωση της κρίσης στην οικονομική κατάσταση των γυναικών και οι δείκτες αυτές πρέπει να αναφερθούν και στα περιβαλλοντολογικά και στα κοινωνικά και στα οικονομικά στοιχεία. Πρέπει να υπάρχει μια συνική παρακολούθηση ε, και μια ε, αναθεώρηση των δικτών οι οποίοι ήδη έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του προγράμματος του Πεκίνου σύμφωνα με ε, τη σχετικότητα του γενικότερου πλαισίου πράγμα το οποίο θα επιτρέψει να υλοποιήσουμε τους κοινούς μας στόχους. Τέλος, μακροπρόθεση πρέπει να υπάρξει μια πολιτική ισότητα ανδρών και γυναικών και μία ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Με αυτή την ε, δομή σε τρία επίπεδα θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους βασικούς μας στόχους. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής έχει ένα λεπτό και είναι η κυρία Ζερία Κώστα. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το Πεκίνο συν 15 αντιμετωπίζει σήμερα μια χρηματοπιστωτική κρίση σοβαρότατη στην Ευρώπη και στον κόσμο που πλήττει κυρίως εκατομμύρια γυναικών αλλά που μπορεί να αποτελέσει όμως και την ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε την οργάνωση της εργασίας, επανοργάνωση των κοινωνικών πολιτικών. Η, Ευρώπη πρέπει να παλέψει για τους στόχους του Πεκίνου ΣΥΝ 15, για τις γυναίκες, για την πρόσβασή τους στις πιστώσεις μέσα από, από τα μικροδάνεια. Θα πρέπει επίσης να προχωρήσει και η οδηγία για την γονική άδεια. Θα πρέπει να προωθηθούν επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέες γυναίκες μία νέα οδηγία για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε την ενίσχυση των γυναικών στις στοχότερες χώρες, πιο συγκεκριμένα στην Αφρική, για να μπορέσουμε με τις γυναίκες να οικοδομήσουμε μία ευρωαφρικανική συμμαχία γυναικών. Θα ήταν καλό εάν η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη ξεκινούσε μία καμπάνια ώστε το Νόμπελ της Ειρήνης να δοθεί στις Αφρικανές γυναίκες, αυτές που παίζουν έναν αρχηγικό ρόλο για την προστασία της ειρήνης στις εμπόλεμες περιοχές. Ευχαριστώ Σιλβία Κώστα. Ένα λεπτό ο επόμενος ομιλητής, η κυρία Γκυγιόμ. Σήμερα συζητάμε για την ισότητα ανδρών και γυναικών και συγχρόνως εορτάζουμε το Ευρωπαϊκό Έτος κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι γυναίκες είναι το πρώτο θύμα της κρίσεως των κακοπληρωμένων και προσωρινών εργασιών ε, κερδίζουν λιγότερο από το κατώτατο επίπεδο αμοιβή ε, και βρίσκονται σε ένα σοβαρό επίπεδο ένδυας. Άρα η ισότητα ανδρών γυναικών είναι περίπου θεωρητική και οι γυναίκες αναλαμβάνουν και τα οικογενειακά βάρη και πρέπει να εργάζονται με ευέλικτα ωράρια και τελικά κερδίζουν λιγότερο. Πρέπει λοιπόν να εξαλειφθούν όλες αυτές οι ανισότητες και να βρούμε μέθοδους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών διαφορετικά οι, διαταγές του, οι επιταγές του Πεκίνου θα παραμείνουν ε, μόνο ένα όνειρο. Το επόμενο ομιλητή είναι ο κύριος Μπλίνκαγε. Η αρχή της ισότητας των δύο φύλων είναι βασική για να επιτύχει η Ένωση Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή. Η Ένωση έχει προοδεύσει στην εφαρμογή της πλατφόρμας του Πεκίνου. Δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι όμως με την παρούσα κατάσταση. Η έκθεση για την εφαρμογή της πλατφόρμας του Πεκίνου δείχνει ότι η Ένωση δεν έχει επιτύχει ακόμα τους στόχους που εθέτονται στο έγγραφο. Οι δείκτες του Πεκίνου πρέπει να παρακολουθηθούν για να παρακολουθήσουμε την ισότητα σε εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στις εκθέσεις για την κοινωνική συμπερίληψη. Ακόμα δεν έχουμε συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα και σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο για να προσδιορίσουμε την φτώχεια των γυναικών ή την βία που πλήττει τις γυναίκες. Θέλουμε συγκρίσιμα δεδομένα για να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα που άπτονται των γυναικών. Οι στόχοι του προγράμματος εργασίας θα προωθήσουν την εξέλιξη των δικτών του Πεκίνου. Τώρα που έχουμε οικονομική κρίση πρέπει να ενισχυθεί η ισότητα των δύο φύλων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπλενκεβετσούτε. Πάμε τώρα στη διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Η κυρία Μαγκίνες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους για τις ε, συνδρομές. Ε, εκπροσωπώ ε, γυναίκες δημοσίου υπαλλήλου, οι οποίες ανησυχούν για το πώς μπορούν να προχωρήσουν πέραν του υψηλού επίπεδου που έχουν επιτύχει. Θα παρακαλούσα τις συναδέλφους στα αριστερά μου να μην γελάνε όταν μιλάω. Με συγχωρείτε κύριοι Βρετανοί φίλοι μου. Με συγχωρείτε δεν είναι πολύ ευχάριστο όταν προσπαθεί κάποιος να μιλήσει και ίσως μπορεί να μην τους ενδιαφέρει αλλά άλλοι ίσως ενδιαφέρονται για αυτά που έχω να πω. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι περνάμε πάρα πολύ χρόνο να προσπαθούμε να προωθήσουμε τις γυναίκες στα επαγγέλματα χωρίς να κοιτάζουμε εάν θα εμπλακούν στα επαγγέλματα αυτά και αυτό λόγω του ότι είναι κακοπληρωμένες. Δεν ε, τις πληρώνουμε αρκετά για να καθαρίζουν χώρου. Ε, και ίσως ας είχαμε μία ισότητα σε αυτό το επίπεδο πριν προχωρήσουμε περαιτέρω και γι' αυτό για να υπάρξει ε, ακριβώς ισότητα των φύλων θα πρέπει να ασχοληθούμε από αυτό το σημείο. Ε, όσον αφορά στη γεωργία και πάλι κάνουν οι γυναίκες πολλές δουλειές οι οποίες δεν υπολογίζονται και αυτό είναι ένα βασικό θέμα των αλλαγών στη γεωργική πολιτική. Δύο άλλα θέματα που θέλω να αναφέρω. Ξέρω ότι πολλές γυναίκες ενεπλάκησαν στη συζήτηση αυτή, αλλά οι γυναίκε έχουν παιδιά. Θα, ε, δεν θα, ε, θα ήμασταν εδώ με τα παιδιά μας. Ε, μπορούμε διότι πληρωνόμαστε πολύ καλύτερα. Εχθέ όμως από τις γυναίκες από το Ιράν ακούσαμε και θα έπρεπε εμεί να αναγνωρίσουμε τον αγώνα τους και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Για ένα λεπτό η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένα βασικό θέμα και εμφανίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διαπιστώσαμε ότι 24% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 33% των αρχηγών των Ευρωπαϊκών ε, ε, ε, επιχειρήσεων ήταν γυναίκες. Ε, ένα μεγάλο ποσοστό νέων γυναικών ε, τουλάχιστον τελειώνει το γυμνάσιο και 50% 50% από αυτούς οι οποίοι τελειώνουν το πανεπιστήμιο θα καλύψουν τις θέσεις εργασίας μέχρι το 2011. Οι γυναίκες όμως έχουν και πολλές μονογονικές ε, οικογένειες όπου μόνο η μητέρα ε, ε, είναι κεφαλή της οικογένειας και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να συμβιβάσουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στους παιδικούς σταθμούς. Παιδικούς σταθμούς για ε, διότι θα πρέπει τα παιδιά τα οποία είναι κάτω των τριών ετών να μπορούν να αποφεληθούν. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Φιγκερέντο. Προέδρε, κυρία Επίτροπε, τώρα που φτάνουμε κοντά στην, στην εκατονταετία της ημέρας των γυναικών και δέκα χρόνια μετά από την έγκριση της πλατφόρμας του Πεκίνιου παρατηρούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή των γυναικών που είναι θύματα της πρόσχερης εργασία, της ανεργίας, της αύξησης των ανισορροπιών, της κρίσης του καπιταλισμού, της βίας στην κοινωνία, στην εργασία και στην οικογένεια. Η φτώχεια είναι θηλυκού γένους, ακόμα και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είναι 85 εκατομμύρια άτομα τα οποία ζουν σε κάτω από το επίπεδο φτώχειας. Υποστηρίζουμε λοιπόν και το ψήφισμα αλλά και εκφράζουμε ότι την ευχή η πλειοψηφία αυτού του κοινοβουλίου να την εγκρίνει και να εγκρίνει και την παράγραφο ότι το αναπαραγωγικό δικαίωμα είναι τμήμα των δικαιωμάτων των γυναικών και είναι απαραίτητο να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για να βελτιωθούν η υγεία των γυναικών και η αναπαραγωγική υγεία των γυναικών στην Ένωση και στον κόσμο και να μην λάβουμε υπόψη στερεότυπα αλλά να προωθήσουμε την ισότητα των δικαιωμάτων ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Η κυρία Κρετού για ένα λεπτό. 95% ε, των γυναιτών προετών ήταν ε, θύματα της βίας. Διαπιστώνουμε όμως ότι ακόμη η κατάσταση δεν έχει διορθωθεί και πολλά προγράμματα απέχουν της πραγματικότητας και οι στόχοι μας δεν έχουν επιτευχθεί. Δυστυχώς όσον αφορά την ε, οικογενειακή βία, τους βιασμούς και ε, την σεξουαλική σκλαβιά ε, όλα αυτά αποτελούν εφιάλτες για τις γυναίκες και αν δεν εμπλακεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη στρατηγική για να αντεπεξέλθουμε όλα τα θέματα τα οποία τελικά καταλήγουν και στην πορνεία ε, διότι η βία δεν είναι για τις γυναίκες αιτία είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να επιλύσουμε Ευχαριστώ και τώρα για ένα λεπτό η, η κυρία Χολμάγερ ο κύριος Χολμάγερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα καλό, ε, μια καλή ένδειξη ότι δεν μιλάνε μόνο οι γυναίκες, διότι η πλατφόρμα του Πεκίνου ε, αποβλέπει στην μη διάκριση. Οι γυναίκες προς ε, την, απέναντι από τους άντρες δεν πρέπει να βρίσκονται σε υποδέστερη θέση. Όσον αφορά την θετική διάκριση ε, θεωρώ ότι ούτε αυτό πρέπει να υπάρχει ε, αντί να ασχολούμαστε όμως με μικροπράγματα θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις πραγματικά καταπιεσμένες γυναίκες που είναι θύματα διακρίσεως που ζουν σε μία παράλληλη κοινωνία και που υφίστανται καθημερινή καταπίεση και βία αφήνουμε μεγάλη ελευθερία στις γυναίκες στην Ευρώπη και αυτό ξεκινά από την ένδυση μέχρι την επιλογή ε, των ε, συζύγων ε, και πού είναι η Ευρώπη των δικαιωμάτων όταν την ψάχνουμε. Υπάρχουν σημαντικές διακρίσεις οι οποίες υπό την κάλυψη της θρησκείας εμφανίζονται καθημερινά και πιστεύω ότι δεν έχουν καμία θέση και πρέπει να καταπολεμηθούν. Ευχαριστώ τον κύριο Μάγερ. Η κυρία Φλασίκοβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν δεν ήταν οι προηγούμενοι ομιλητές, μόνο εμείς γυναίκες και η κυρία Επίτροπος θα συζητούσαμε για αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά είναι ένα επίγον θέμα για την μοντέρνα κοινωνία και συμφωνώ και με τους συναδέλφους, πρέπει να συντονίσουμε τις δραστηριότητες μας σε όλα τα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν της ανισότητας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, βλέπουμε ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερους δείκτες για την αξιολόγηση της ισότητας. Θα πρέπει η Κομισιόν να ζητήσει από την Eurostat να βελτιώσει την, το συντονισμό για την συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων από τα κράτη-μέλη και να καλέσει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με την Eurostat. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων και έχουμε καλές εμπειρίες με τις οποίες, μπορούμε, τις οποίες μπορούμε να μοιραστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο και να τις διαβιβάσουμε περαιτέρω. Και νομίζω ότι σε πέντε χρόνια καιρό όταν θα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια από την πλατφόρα του Πεκίνου, θα έχουμε προοδεύσει περισσότερο. Κυρία Χωρίς μικρόφωνο. Η ισότητα των φύλων είναι μια ουσιαστική αρχή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται και στις συνθήκες και στα πρωτοσέλιδα. Και ε, πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί συζητάμε συνέχεια το θέμα αυτό, διότι σε πάρα πολλούς τομείς δεν υπάρχει ισότητα. Και προσβλέπω στην ημέρα που δεν θα χρειάζεται πλέον να μιλάμε για την ισότητα των φύλων ε, στο κοινωνικό βίο, διότι θα έχει καταστεί πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπες Γκαρίδα, ξενόμενο του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημερίζομαι όλες τις τοποθετήσεις των ομιλητριών. Όλες ήταν ομιλήτριες εκτός από τον κύριο Όμπερ του οποίου όμως την τοποθέτηση μερικώς συμμερίζομαι. Πρέπει να πω ότι αυτές οι τοποθετήσεις των κυριών αποτελούν έκφραση αυτής της νέας φάσης που ξεκινάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα των φύλων. Η ισότητα των φύλων που δεν ευεργετεί μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Η ισότητα των φίλων... είναι μια ουσιαστική αρχή στάθμισης. Γι' αυτό εγώ φανταζόμουν ότι σήμερα θα τοποθετιόντουσαν τόσες όσες γυναίκες όσοι και άντρες. Γιατί για όλους μας είναι καλό, όχι μόνο για τις γυναίκες. Εγώ πιστεύω ότι πολύ σωστά στο άρθρο 2 της Ένωσης για πρώτη φορά στα πλαίσια πρωτογενούς δικαίου μιλάμε για ισότητα των φύλων και στο άρθρο 8 της θήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέμε ότι όλες οι πολιτικές θα πρέπει να διέπονται από την ισότητα των φύλων. Πρόκειται λοιπόν για τον πυρήνα της άσκησης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο τώρα θα κάνουμε στην πράξη είναι να εφαρμόσουμε αυτή την εντολή που μας δίνει η συνθήκη. Αυτό το οποίο θέλει να κάνει το Συμβούλιο της Ένωσης και η Ισπανική Προεδρία. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και τη συνεργασία της Κομισιόν. Ε, Χθε είχαμε μια συνεδρία στη Μαδρίτη, ήταν παρούσα η Επίτροπος, η κυρία Ρέντιν και θα έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με την Κομισιόν, ούτω ώστε οι φιλοδοξίες μας για την ισότητα των φύλων θα γίνουν πραγματικότητα σε αυτή την Προεδρία. Και για να μιλήσω για το εγκύτερο γεγονός, θα αναφερθώ στις 8 Μαρτίου. Στις 8 Μαρτίου όπου το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο θα συζητήσει τη χάρτα των γυναικών και το Συμβούλιο θα συζητήσει το θέμα της εγκρίζωσης της βίας κατά των γυναικών. Η βία μεταξύ των φίλων είναι η χειρότερη μάστιγα στις κοινωνίες μας. Το χειρότερο στην κοινωνία μας είναι η βία κατά των γυναικών και η εξάλληψή της θα είναι πραγματικά μία κατάκτηση. Γιατί ως κατάκτηση θα πρέπει να το ρίσουμε για τους επόμενους μήνες. Τόσο της Κομισιόν όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Λόπες Γκαρίδο εξ ονόματος της Επιτροπής η κυρία Ρέντινγκ. Πρόεδρε, οι οδηγίες περί ισότητας ξεκίνησαν τη δεκαετία του 70 και έκτοτε πολλές οδηγίες έχουν όχι μόνο αλλάξει την νομοθεσία των κρατών μελών, αλλά τους δημιούργησαν γιατί δεν υπήρχαν τότε νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Η νομοθεσία για ισότητα μεταξύ άντρες και γυναίκες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας μας. Και παρόλα αυτά, και έχετε δίκιο σε αυτό, βλέπετε ότι έχουμε καλούς νόμους, όμως η πρακτική δεν τους ακολουθεί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι όχι να δημιουργήσουμε νέους νόμους, αλλά να φροντίσουμε ώστε να εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι στην κοινωνία. Εγώ ονειρεύομαι μια στιγμή όταν θα κάνουμε μια συζήτηση εδώ και το 50% των γυναικών και το 50% των ανδρών θα είναι ομιλητές. Ονειρεύομαι να μην χρειαζόμαστε πλέον την Διεθνή ημέρα της γυναίκας διότι δεν θα υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα. Όμως καλά να κάνει κανένας να ονειρεύεται, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Γι' αυτό λοιπόν και είμαι ευγνώμων την Ισπανική Προεδρία που έβαλε το θέμα των γυναικών ως προτεραιότητά της και είμαι αποφασισμένη μαζί με τους συναδέλφους μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ενσωμάτωση της ισότητας ανδρών και γυναικών να μπει σε όλες τις πολιτικές που θα σας παρουσιάσουμε. Και παρεπιπτόντος, μαζί με τον συνάδελφο κύριο Άντορ που είναι υπεύθυνο για θέματα απασχόλησης, θα φροντίσουμε στην, στο πρόγραμμα για το 2020 και αυτό να συμπεριληφθεί για τα υπόλοιπα στοιχεία. Όπως έχω ήδη πει, θα συνεργαστώ με τις οργανώσεις των γυναικών για την νέα στρατηγική για την ισότητα όπου θέματα οι γυναίκες σε θέσεις υπευθυνότητας θα είναι προτεραιότητα γιατί αυτά είναι διαρθρωτικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν και θέματα που αφορούν την ίδια την κοινωνία και τα οποία είναι πολύ βαθιά και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την βοήθεια των οργανώσεων γυναικών, με την βοήθεια των υπουργών στα κράτη-μέλη, με την βοήθεια των εθνικών νόμων, με την βοήθεια των ευρωπαϊκών νόμων. Και αυτό είναι το τρομερό θέμα της βιαιότητας κατά των, της βίας κατά των γυναικών. Νομίζω ότι αυτά θα είναι στο προσκήνιο των εργασιών που θα κάνουμε και νομίζω ότι παρόλα αυτά κυρίες μου όταν η ισχυρή σας αντιπροσωπεία θα πάει στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει τα 15 χρόνια της πλατφόρμας του Πεκίνου. Νομίζω ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, διότι αν δούμε τι έχουμε πετύχει στα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε πετύχει πολλά. Δεν έχουμε βεβαίως φτάσει εκεί που ονειραβόμασταν ότι θα έχουμε φτάσει, όμως έχουμε πετύχει πολλά και μέσω αυτής της εμπειρίας μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε και τις γυναίκες σε άλλες υπήρους. Και αυτό θα είναι το αντικείμενο της συνάντησης στη Νέα Υόρκη. Όχι μόνο να δούμε τι κάνουν οι Ευρωπαίες γυναίκες, αλλά τι οι Ευρωπαίες γυναίκες και οι ευρωπαϊκές πολιτικές, οι αναπτυξιακές πολιτικές της Ευρώπης μπορούν να κάνουν για τις γυναίκες της άλλες υπήρους. Και πιστεύω ότι η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι ένα πολύ όμορφο κείμενο το οποίο θα πρέπει να αναγνώσει κάθε παιδί σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία. Θα πρέπει να το έχει επεξεργαστεί κάθε φοιτητή στα πανεπιστήμια μας. Αυτός λοιπόν ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων πραγματικά τονίζει τα πράγματα όπως είναι. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα, είναι ίση και είναι ευθύνη μας να φροντίσουμε όταν δεν εφαρμόζεται στην νομοθεσία μας τα κράτη-μέλη αυτή η βασική αρχή να διαμαρτυρόμαστε. Δεν πρέπει μόνο να το κάνουμε εδώ αλλά και στα κράτη-μέλη μας και να δείχνουμε τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν και τα οποία δεν επιλύονται και όχι να σιωπήσουμε και θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους τους άνδρες σε αυτό το κοινοβούλιο και εσείς να φωνάξετε μαζί με τις γυναίκες. Ξέρετε ότι το Προεδρείο δεν μπορεί να σχολιάσει, οπότε θα πω από σχόλια. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό το σημείο και αύριο στις 11.30 θα ψηφίσουμε το σχετικό ψήφισμα. Πάμε τώρα στις τοποθετήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 150. Είναι η τοποθετήση ενός λεπτού. Και θα έχουν την προτίμηση